Um, Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Να ξεκινήσουμε τη συνάντησή μας. Η κυρία Γκρέστερ θα είναι μαζί μας σύντομα, αλλά μπορούμε να ξεκινήσουμε με τις ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Να ξεκινήσουμε με κάτι ευχάριστο. Είναι τα γενέθλια της Μπέρκη Σίπελ. Είναι ο πιο ωραίος τρόπος να ξεκινάει η συνεδρίαση. Χρόνια πολλά, Μπέργη, και ό,τι καλύτερο. Και θα περάσεις αυτή τη μέρα στην Επιτροπή Λίμπε με τους φίλους σου. Ελπίζω να περάσει όμορφα σήμερα. Σου εύχομαι λοιπόν ό,τι καλύτερο για τα γενέθλιά σου. Λοιπόν, εγκρίνουμε την ημέρα διάταξη, συνάδελφοι. Υπάρχει μια αλλαγή στο σχέδιο ημέρα διάταξη, στο σημείο 5α, αναφορά στην Επιτροπή για τις διαπραγματεύσει σχετικά με τις θεωρήσεις θα γίνει στις 15.35 και στο σημείο 9 ε, Eurojust και Γεωργία 4 Φεβρουαρίου τελικά θα εξεταστεί αυτό και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις αυτή είναι και η τροποποιημένη ημερήσια διάταξη τα ε, πρακτικά της συνδρίας της 5ης Μαρτίου έως τις, καθώς και στις 15 Οκτωβρίου και στις 8 Νοεμβρίου ε, εγκρίνονται εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις Τώρα για το γλωσσικό καθεστώς υπάρχει σήμερα διερμηνία σε όλες τις γλώσσες εκτός από δανικά, κροατικά και ιρλανδικά. Έχουμε και άλλες ε, πράξεις δεξιόδότηση και ε, εφαρμοστικές πράξεις οπότε παρακαλώ πρέπει να παρακολουθήσετε για τις πράξεις ε, από μια πολιτική ομάδα έχει υποβληθεί αντίρρηση για έναν από τους κανονισμούς ε, εξιοδότησης. Οι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες 18 Δεκεμβρίου μας στείλαν την ε, αντίρρησή τους. Έχει να κάνει με το ε, Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, Εξωτερικά Σύνορα και Θεωρήσεις, καθώς και για το άσυλο, τη μετανάστευση και την ένταξη, το σχετικό ταμείο δηλαδή. Υπάρχουν λοιπόν δύο, έχουν αποσταλεί δύο σχέδια αντιρρήσεων στην γραμματεία της ΛΥΜΠΕ έχουν υποβληθεί προς απόφαση σήμερα, στη σημερινή συνεδρία των συντονιστών που θα λάβει η χώρα σήμερα στο τέλος της συνάντησής μας. Για τα εφαρμοστικέ πράξεις, 23 Ιανουαρίου το Κοινοβούλιο έλαβε δύο παραρτήματα στην, στο σχέδιο εφαρμοστικής απόφασης της Κομισιόν που εγκρίνει την τρίτη αναθεώρηση του σχέδιου εργασιών που εφαρμόζει το πρόγραμμα για τη διαλειτουργικότητα και το κοινό πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Δημοσίων Υπηρεσιών ε, επιχειρήσεων και πολιτών, το πρόγραμμα ΙΣΑ, καθώς και οι δαπάνες, οι δημοσιονομικές σχετικές για το 2019. Βασιζόμαστε ε, στη βασική πράξη, στην απόφαση 2015-2240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με ημερομηνία 25 Νοεμβρίου 2015, που θεσπίζει ένα πρόγραμμα για λύσεις διατουργικότητας ε, και κοινά πλαίσια σε ό,τι αφορά τι ευρωπαϊκέ δημόσιε υπηρεσίε, ε, τι επιχειρήσει και του πολίτε ε, για τον εξυγχρονισμό του δημόσιου τομέα. Αυτά τα παραρτήματα έχουν αποσταλεί σε όλα τα μέλη της ΛΥΜΠΕ μέσω του newsletter στις 25 Ιανουαρίου 2019. Αν ένα μέλος έχει αντιρρήσει, ε, παρακαλώ να ενημερώσει την γραμματεία της ΛΥΜΠΕ πριν τις 6 Φεβρουαρίου 2019 στις 12 το μεσημέρι. Okay, so, um, for the next item... Το, το πρώτο σημείο που θα μας απασχολήσει σήμερα, ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκινούμε τον πρόεδρο της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου η οποία όμως δεν έχει έρθει ακόμα ξέρει βεβαίω όσοι γνωρίζουν την κυρία Γκρέτσερ ξέρουν ότι είναι εξαιρετικά ακριβή και επειδή είναι ακριβή, περιμένουμε ακόμα λίγο. Επειδή λοιπόν είναι ακριβή, θα διακόψουμε για λίγο. There is no, there is no on my Ε, δεν είναι ότι χαίρομαι εδώ ε, με, τα, προβλήματα των άλλων. Δεν είμαι χερέκακος. Πάντα ε, μου αρέσει να συμπροεδρεύω με την κυρία Γκρέσλερ, οπότε θα περιμένουμε λίγο ακόμα. Φτάνει. Φτάνει, έρχεται. Ε, οπότε περιμένετε ακόμα, περιμένουμε ακόμα λίγα λεπτά. pause for maybe one minute and uh, Mrs. will be with us. Thank you. Okay, thank you, colleagues, and... Uh, Ευχαριστώ συνάδελφοι. Ήρθε λοιπόν η κυρία Γκρέσλερ και μπορούμε να ξεκινήσουμε. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Όλιβερ Σάλες που ε, ορίστηκε τον περασμένο Οκτώβρη ως ενδιάμεσος διοικητικός, ε, διε, ναι, διοικητικός διευθυντής της ΕΠΟ, της Ευρωπαϊκής Αγγελία, σύμφωνα με τον κανονισμό 2017-1939 που θεσπίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο κ. Άλλη παίζει ένα πολύ κρίσιμο ρόλο στον καθορισμό και την αρχική επιχείρηση, ε, ε, ε, αρχική λειτουργία της ΕΠΟ. Είμαι πεπισμένο ότι θα μας δώσει μια σαφή εικόνα της προπαρασκευή που έχει να κάνει με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είμαστε στη φάση της ε, λειτουργίας πλέον της ΕΠΟ και βεβαίως υπάρχει διαδικασία για τον ορισμό του Ευρωπαίου Γενικού Εισαγγελέα. Ε, θα δώσω τώρα το λόγο στη συνάδελφο, την κυρία Γκρέσλε, ε, μιας και έχουμε κοινή συνάντηση της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου. Ε, έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Κλοντ. Ε, συνάδελφοι, ζητώ συγγνώμη που άργησα. Είχα όμως κάποιους δημοσιογράφους και δυστυχώς ε, δεν εξαρτηθόταν από μένα. Λοιπόν, είναι σημαντικό αυτό το θέμα για μας. Έχουμε εναποθέσει μεγάλες ελπίδες ε, σε αυτήν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γι' αυτό και θέλω να συμφωνήσουμε εδώ, να ορίσουμε κοινέ ημερομηνίε για να γίνουν οι ακροάσει. Και βεβαίω να εξασφαλίσουμε ότι η Κομισιόν θα μα ενημερώσει έγκαιρα ε, σε ποιο σημείο βρίσκεται όσον αφορά την ε, θέσπιση αυτή τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πώς τελικά υλοποιείται αυτό το σχέδιο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει αυτόν τον, ε, αυτήν την εισαγγελία και να στελεχωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτύχουμε γρήγορα ε, και πολύ θετικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ, Ίγκε. Ε, να δώσω το λόγο στον κύριο Σαλ. Σας καλωσορίζω. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ και χαίρομαι για την ευκαιρία για να, που έχουμε να κάνουμε σήμερα αυτή την ε, κοινή συζήτηση με τις δύο επιτροπές σας. Είναι η πρώτη μας ευκαιρία, αλλά φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν ε, και επόμενες ευκαιρίες στο μέλλον για να σας ενημερώνω. Ε, εγώ λοιπόν διορίστην τον προηγούμενο Νοέμβριο από την Κομισιόν ως προσωρινός διευθυντής ε, νομίζω ότι κομίζω αρκετή εμπειρία. Εργάζομαι στην Κομισιόν εδώ και 25 χρόνια και ε, έχω ασχοληθεί με ζητήματα δημοσιονομικά, ανθρώπινων πόρων, αλλά και με την δημιουργία άλλων φορέων, όπως ε, το Single Resolution Board, στο παρελθόν. Πρόθεσή μου είναι να σας ενημερώσω για το πού βρισκόμαστε όσον αφορά την θέσπιση και την προπαρασκευαστική φάση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και συγκεκριμένα του, την επιλογή του επικεφαλής της και στη συνέχεια βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Προφανώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της κατασκευής, της προετοιμασίας της και σε αυτή τη φάση προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε διάφορες ε, δομικές μονάδες. Κάποιες είναι πολύ συγκεκριμένες, να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Για παράδειγμα, ε, συνεργαζόμαστε στενά με τις λουξεμβουριανές ε, αρχές για το κτίριο οι λουξεμβουργιανές αρχές δηλαδή μας έχουν ε, προτείνει ένα συγκεκριμένο ε, κτίριο στο οποίο γίνονται κάποιες τελευταίες εργασίες αυτή τη στιγμή ε, και θα είναι στη διάθεσή μας στις αρχές του 2020. Είναι ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό, αποδοτικό και ασφαλές κτίριο. Επίσης, ε, εργαζόμαστε επί ενός συστήματος διαχείρισης ε, υποθέσεων που θα συνδέει τις διάφορες αρχές αλλά θα ευκολύνει και την ανταλλαγή και διαβίβαση δεδομένων και πληροφοριών που σχετίζονται με τις υποθέσεις και ε, στο, στον τομέα αυτό έχουμε ζητήσει και την... Έχουμε ζητήσει και την βοήθεια διαφόρων εξωτερικών εμπειρογνωμόνων ε, έχουμε επίση έρθει σε επαφή με διάφορου φορεί, ε, Eurojust, Europol, την ε, Γενική Διεύθυνση δικαιοσύνη, τον Όλαφ και εκπονούμε και μια σχετική μελέτη, τα πορίσματα της οποίας θα δημοσιευθούν τον Μάρτιο και από εκεί και πέρα θα συζητήσουμε και με τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο της ομάδας εμπειρογνωμόνων για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Άλλοι τομείς στους οποίους σημειώνουμε πρόοδο είναι ε, ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που εγκρίθηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2019 και εδώ θέλω να ευχαριστήσω ε, και το Κοινοβούλιο για τη συμβολή του. Έχουμε έναν προϋπολογισμό 4,9 εκατομμύριων ε, ευρώ που θα μας επιτρέψει να ξεκινήσουμε αυτή την πρώτη φάση λειτουργίας αυτού του νέου φορέα μηχανογραφικά συστήματα, προσλήψεις προσωπικού και είμαστε βέβαιοι ότι τα πράγματα θα έχουν θετική έκβαση την πρώτη χρονιά ε, των επιχειρήσεων. Θα δούμε βεβαίως και στην ενδιάμεση περίοδο αν θα αρκέσει ο συγκεκριμένος προπολογισμό, αλλά αυτό μένει να αποδειχθεί. Το σημαντικότερο βεβαίως, ε, το οποίο δεν σας έχω πει ακόμα, είναι ο διορισμός του επικεφαλής. Ξέρετε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις στον ιδρυτικό κανονισμό και συγκεκριμένα όσον αφορά τον διορισμό, την επιλογή μάλλον και τον διορισμό τόσο του, ε, της Επιτροπής Επιλογής ε, στην οποία συμμετέχει και ένα μέλος το οποίο προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πού βρισκόμαστε τώρα όσον αφορά την επιλογή του επικεφαλής. Οι εργασίες αυτές ξεκίνησαν ήδη τον Νοέμβριο και η πρώτη συνάντηση αυτής της Επιτροπής Επιλογής έγινε πριν τα Χριστούγεννα, όπου και επικεντρωθήκαμε σε πρακτικά επιχειρησιακά ζητήματα, για να καταρτήσουμε ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα το οποίο θα, δώσει, θα έδινε στη δυνατότητα και στην Επιτροπή αλλά και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να ασκήσουν τις αρμοδιότητες τους και τον ρόλο τους σωστά. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων, τα μέλη αυτής της Επιτροπής Επιλογής ανέλησαν σε βάθος όλες τις αιτήσει που παρελήφθησαν και αυτό τους έδωσε τη δυνατότητα να ε, πραγματοποιήσουν τον Ιανουάριο μια αγώνιμη ε, συνάντηση όπου και καταρτίστηκε ένας ε, περιορισμένος κατάλογος 11 υποψηφίων για συνέντευξη. Και αυτές οι συνεντεύξεις θα γίνουν αύριο και μεθαύριο. Η Επιτροπή Επιλογής λοιπόν ελπίζει βάσιμα ότι θα μπορέσει να διαβιβάσει αυτόν τον σύντομο κατάλογο υποψηφίων ε, σε δύο εβδομάδες στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Στους εφαρμοστικούς κανόνες του Συμβουλίου ορίζεται ότι στόχος είναι να καταλήξουμε σε τρεις έως πέντε υποψηφίους και αυτό θα εξαρτηθεί βεβαίως από το τι θα προκύψει από τις συνεντεύξεις που θα γίνουν τις επόμενες μέρες. Ελπίζουμε όμως ότι η Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού θα καταφέρει να επιλέξει και να προσδιορίσει τους πλέον κατάλληλους υποψηφίους και να τους θέσει στη συνέχεια υπόψη του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Στο σημείο αυτό θέλω να τονίσω ότι για την ορθή λειτουργία της Ευρωπαϊκής εισαγγελία είναι πολύ σημαντικό τα δύο θεσμικά όργανα να ακολουθήσουν τα απαραίτητα βήματα, τα οργανωτικά για τις ακροάσεις, ώστε να καταφέρουμε να προτείνουμε και στη συνέχεια να διορίσουμε τον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής εισαγγελία πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές και ελπίζουμε δε στην τελευταία ολομέλεια του Κοινοβουλίου τον Μάρτιο. Και για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται καλός συντονισμός ώστε να εξασφαλίσουμε ότι όλο το χρονοδιάγραμμα θα τηρηθεί. Και επίσης να σας ενημερώσω σχετικά με την επιλογή των άλλων μελών του κολογίου, των Ευρωπαίων Εισαγγελέων δηλαδή, που πλέον θα είναι 22 μετά τις, την προσθήκη των, ε, της Μάλτας και των κάτω χωρών και όχι 20. Οι κύριοι Γιούροβα και ε, Έτιγκερ ε, συναντήθηκαν το Δεκέμβριο με όλους τους αρμόδιους εθνικούς υπουργούς ζητώντας τους να ξεκινήσει η εθνική διαδικασία επιλογής και ζητώντας τους να υποβάλουν εκείνη τις προτάσεις τους τριών ονομάτων έως τα τέλη Μαρτίου. Το χρονοδιάγραμμα λοιπόν είναι ότι θα λάβουμε τις προτάσεις και από τα 22 κράτη-μέλη έως τα τέλη του Μαρτίου και από εκεί και πέρα η Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού θα αρχίσει, να ξεκινά, θα αρχίσει την ε, δεύτερη φάση της εντολής της, δηλαδή τον έλεγχο, ε, την εξέταση και τη δημιουργία, ε, την πραγματοποίηση συνεντεύξεων με τους προτινόμενους υποψηφίους από τα κράτη-μέλη, ώστε στη συνέχεια να μπορεί η Επιτροπή αυτή να διαβιβάσει τις προτάσεις της στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο λίγο αργότερα. Δεν έχουμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ακόμη αυτή τη στιγμή, αλλά θα προσπαθήσουμε το συντομότερο δυνατό και σε συνεργασία με τις διάφορες γραμματείες να το καταρτήσουμε. Και τέλος, επιτρέψτε μου επίσης να σας πω ότι πριν από λίγες μέρες, στις 11 Ιανουαρίου, η Κομισιόν υπέβαλε ε, σχέδιο πρότασης για εφαρμοστική απόφαση του Συμβουλίου όσον αφορά τους μεταβατικούς κανόνες για το διορισμό των ε, πρώτων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Γιατί προφανώς ε, στην πρώτη φάση της εντολής αυτής θα πρέπει να βρεθεί μια μεταβατική προσωρινή λύση. Αυτά είχα να σας πω. Η δουλειά αυτή προχωρά σταδιακά, υπάρχουν πλέον κάποια απτά αποτελέσματα ε, πρέπει τώρα η Κομισιόν να διαχειριστεί τις ροές εργασιών που επίκυνται να ολοκληρωθούν ε, το επόμενο διάστημα και ελπίζουμε τους επόμενους μήνες να καταφέρουμε να, καταρτήσουμε και να ε, θέσουμε σε λειτουργία τη νέα Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ευχαριστούμε πολύ. Θα κοιτάξουμε σύντομα τον κατάλογο των υποψηφίων, το δεύτερο μέρος Πολλοί συνάδελφοι εδώ νομίζω ενδιαφέρονται θερμά για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Παρακαλώ, όποιο θέλει, έχει το λόγο για κάνα δίλεπτο καθένα. Κυρία Μετσόλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, εντάχει, θα ήθελα να εκφράσω την πλήρη μου υποστήριξη για την για τον άμεσο διορισμό του επικεφαλής στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Διαρκώς ακούμε για έρευνες ε, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το πώς γίνεται κατά ε, εξαίρεση κακή κακοδιαχείριση των σχετικών κονδυλίων. Πρέπει λοιπόν να αποστείλουμε ένα σαφές μήνυμα. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να δώσουμε τις κατάλληλες απαντήσεις. Απαντήσεις που να έχουν και κάποιο νόημα για την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Ωστόσο, οι κανόνες για το πώς θα ε, επιλεγούν οι υποψήφοι και θα γίνουν οι διορισμοί είναι ένα θέμα διαδικαστικό. Και βεβαίως ε, επηρεάζεται και από τις επικείμενες ευρωεκλογέ. Ε, τα διαδικαστικά ζητήματα και οι αποφάσεις για τους διορισμούς, επειδή είναι ιδιαίτερα λεπτής φύσης, θα μπορούσαν να συζητηθούν σε συνεδρία σε συντονιστών πιστεύω εγώ, όπου θα εκπροσωπούνται όμως όλες οι πολιτικές ομάδες και θα μπορούμε να προχωρήσουμε αμέσως ώστε οι διορισμοί να γίνουν εντός του διαστήματος της θητείας μας. Ευχαριστούμε Ρομπέρτα. Από την Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών, η κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστώ και τον κύριο Σάλ για την ενημέρωση. Έχουμε φτάσει πλέον στα 22 κράτη-μέλη που συμμετέχουν ε, στην προπαρασκευή πλέον της υποψηφιότητα. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν λάβατε υπόψη σας διότι ξέρετε ότι είναι ένα θέμα που μας πασχόλει σε επίπεδο δημοσιονομικού ελέγχου το λέμε για κάθε υποψηφιότητα Εάν λοιπόν λάβατε υπόψη ε, την ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων σε ό,τι αφορά τη σύνθεση της αγγελίας. Διότι στον, στον τομέα ε, των, της νομικής ε, υπάρχει και η ψηλότερη συμμετοχή των γυναικών. Όμως ε, στο πολύ υψηλό επίπεδο δεν, είναι, δεν υπάρχει ισορροπία Οπότε βεβαίως ο εισαγγελέας πρέπει να έχει μεγάλη εμπειρία και συνήθως ε, αγνοούμε κάποιες γυναίκες εισαγγελείς με μακρά εμπειρία και που έχουν και μια ευρωπαϊκή προσέγγιση συχνά. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα τους πόρους που θα έχει στη διάθεσή του ο νέος εισαγγελέα. Ε. Πού βρισκόμαστε. Οι ανθρώπινοι πόροι, οι διοικητικοί πόροι, ε, τι θα βρει ο άνθρωπος αυτός για να δουλέψει αφού οριστεί. Διότι και από αυτού είναι σημαντικό να δώσουμε κάποιες εγγύησεις, να δώσουμε κάποια ασφάλεια ε, σε αυτόν τον νέο θεσμό, κάποια χέγγια. Μέσω της πρότασης της κυρίας Γκρέσλε λοιπόν, στα πλαίσια του οικονομισμού Όλαφ, θα μπορούσαμε εντός των επόμενων μηνών να φροντίσουμε να προχωρήσουν παράλληλα αυτά για να μην προκύψουν προβλήματα στη μετάβαση από τη μία οργάνωση στην άλλη, να υπάρξει δηλαδή συνεργασία και να μην έχουμε επικαλύψεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Ινές Μπέργκη Τσίπελ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε και ευχαριστούμε και για τις ωραίες σας ευχές για τα γενεθλιά μου σήμερα. Ε, εδώ νομίζω είναι ενδιαφέρον εδώ στο Κοινοβούλιο να υπογραμμίσουμε τη σημασία της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Εισαγγελίας διότι το Κοινοβούλιο ανέκαθεν υπήρξε υπέρ αυτής της ιδέας όχι μόνο για να προστατεύουμε τα οικονομικά και δημοσιονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωση, αλλά ταυτόχρονα να πρασπιστούμε και τα συμφέροντα των φορολογουμένων μας, των απλών πολιτών. Ταυτόχρονα όμως τώρα κάνουμε λόγο για την Ευρωπαϊκή Δημόσια Εισαγγελία Οπότε πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ο νέος αυτός θεσμός θα είναι πλέον αποτελεσματικός ε, ε, στα καθήκοντα που θα αναλάβει ενώπιον των πολιτών μας. Και κυρίως ό,τι αφορά το ποινικό δίκαιο και τις ποινικέ έρευνες. Ε, δεν μπορώ λοιπόν παρά να επαναλάβω αυτό που υπόθηκε και Σήμερα το βράδυ θα έχουμε συνεδρίαση συντονιστών ε, της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, ήδη, οπότε καλό θα ήταν να έχουμε εκεί μια πρώτη ανταλλαγή για να δούμε ποια είναι η σωστή διαδικασία για την επιλογή του καλύτερου υποψηφίου του πλέον λαμπρού για να ξεκινήσει αμέσως τη δουλειά του στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και μετά θα παρουσιάσουμε τι προτάσει μα σε ολόκληρη την Επιτροπή, ώστε να περάσουμε και σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Αλλά θα ξεκινήσουμε, νομίζω, με τη συνεδρία των συντονιστών, συνεδρία των και θα καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα ήδη απόψε. Ευχαριστούμε, Μπίργκιτ. Ναταλή, θέλει το λόγο. Ευχαριστώ, Κλοντ. Απλώς να εκφράσω και εγώ την ικανοποίησή μου για όσα μας είπατε περί διαδικασίας. Περιμένουμε με ανυπομονησία να δούμε το προφίλ των υποψηφίων στον κατάλογο. Είμαστε πολύ κοντά στο στόχο. Και ε, Όπω πολλοί από εμά είπαμε ήδη, συμμερίζομαι και εγώ το γεγονό ότι τώρα που πρέπει να δούμε πώ θα διαμορφωθεί το αρχιτεκτόνημα, θα πρέπει να σκεφτούμε και πώ μπορεί να επεκταθούν οι αρμοδιότητε τη Αγγελία. Αυτό το συζητήσαμε και την περασμένη εβδομάδα όταν η Ρουμανική Προεδρία ε, παρουσίασε τι προτεραιότητέ τη στην Επιτροπή μα. Να δούμε κατά πόσο μπορεί να επεκτείνει τι αρμοδιότητε τη Αγγελία για την καταπολέμηση και τη τρομοκρατία. Να υποφεληθούμε από αυτό τον νέο θεσμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Ναταλή. Η κυρία Ζολή. και εγώ ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, ασκόντα καθήκοντα εκτελεστικού διευθυντού του κύριο Σάλ Χαίρομαι πολύ που έχουμε φτάσει στο στάδιο επιλογής υποψηφίων ήδη του επικεφαλής δηλαδή της εισαγγελίας. Απλώς κάπως ανησυχώ γιατί οι εισαγγελίε που θα προταθούν από τα κράτη αρχικά θα είναι τρεις από, το από την κάθε χώρα. Ε, έχουμε προβλέψει η επιτροπή που θα κάνει την επιλογή να μπορεί να ελέγξει και το βιογραφικό και την ποιότητα των υποψηφίων για χώρες όπως η Πολωνία, η Ρουμανία, που δεν σέβονται και πολύ το δικαστικό σύστημα ίσως να μπουν στον πειρασμό, να μας στείλουν εισαγγελείς αφού κάπως ε, παραμερίσουν κάποιους καταλληλότερους. Ποιος λοιπόν θα ελέγχει την ποιότητα των ε, εισαγγελέων των ερευνητών ανακριτών και όχι μόνο των γενικών εισαγγελέων. Ευχαριστούμε κυρία Ζολή. Θέλετε να απαντήσετε κύριε Σάλ. Α, μισό λεπτό. Κυρία Μακοβέη. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ καλώς ορίζω ε, την προβλεπόμενη συνεδρίαση των συντονιστών, γιατί κάποια πράγματα πρέπει να αποσαφανιστούν, ιδίω ω προ τη διαδικασία για την σωστή επιλογή, τον εντοπισμό τέλο πάντων του πώ θα πρέπει να επιλεγούν υποψήφοι σε κάθε κράτο μέλο για τους γενικούς εισαγγελίους. Και ως προς τον προπολογισμό, δεδομένου ότι τώρα σε κάθε κράτο μέλο θα προταθούν δύο αρμόδιοι εισαγγελεί. Μπορεί για κάποια κρατημέλη αυτά που προτείνονται στον προπολογισμό να μην είναι αρκετά. Μήπω θα μπορούσαμε να προβλέψουμε ο προπολογισμό του 2020 να καλύψει τα κενά ε, με μια αύξηση. Δεν θέλω να δώσω παραδείγματα συγκεκριμένων χωρών, αλλά μιλάμε για χώρε όπου η διαφθορά σοβεί. Τέλος, να ευχαριστήσω τον κύριο Σάλ για τη δουλειά του και να πω ότι οι διορισμοί καλό θα να γίνουν όσο το δυνατόν συντομότερα. Συμφωνώ με τη Ρομπέρτα απολύτω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Μακοβέη, οπότε κύριε Σάλ, παρακαλώ απαντήστε. Merci, Monsieur le Président, et merci aux, différents membres Ευχαριστώ Πρόεδρε και να ευχαριστήσω και τα μέλη του Κοινοβουλίου που με υποστήριξαν, που μας υποστηρίζουν. Είναι κάτι που το εκτιμούμε. Να απαντήσω δύο-τρία επιμέρους θέματα τα οποία τέθηκαν. Πρώτα απ' όλα για να απαντήσω στην κυρία Σάντερς, για το, την κυρία Σέντερ για τα ζητήματα ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Βεβαίως και είναι ε, σημαντικό αυτό και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τα μέλη του πάνελ επιλογής η Κομισιόν ε, είχε βεβαίως εδώ ένα, ε, μια εξουσία, αν μια αρμοδιότητα ε, στην επιλογή του πάνελ. Πέντε από τα δώδεκα μέλη είναι γυναίκες του πάνελ επιλογής και εργαζόμαστε σε απόλυτη αρμονία με όλα τα μέλη του πάνελ και με αυτές τις πέντε γυναίκες. Τώρα, βεβαίω, οι υποψηφιότητε για την εισαγγελία δεν εξαρτώνται από εμά. Πάντω, υπήρχαν πολλέ γυναίκε μεταξύ των 30 υποψηφιότητων που λάβαμε και πολλές γυναίκες επίσης ε, ε, θα περάσουν από τις συνεντεύξεις αύριο και μεθαύριο μεταξύ των 11. Θα εξαρτηθεί βέβαια και από την ποιότητα, το πώς θα πάνε στις συνεντεύξεις, ε, έτσι ώστε να έχουμε γυναίκες στον, στην τελική short list. Εγώ θα το ήθελα αυτό. Καλό είναι να υπάρχει ισορροπία και στον τελικό κατάλογο. Και κάτι ακόμα για τη μελλοντική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Βεβαίως, όταν ο επικεφαλής, ο Γενικός Εισαγγελέας θα αναλάβει τα καθήκοντά του, είτε αυτό γίνεται το καλοκαίρι, λίγο πριν, λίγο μετά, ε, θα έχει στη διάθεσή του μία ομάδα ατόμων, μία μικρή ομάδα καταρχήν της Κομισιόν, συνάδελφοι από την Όλα, την Γενική Διεύθυνση ε, αυτή τη στιγμή προσλαμβάνουμε και κάποιου ανθρώπου που θα μπορούν να βοηθήσουν σε διοικητικό αλλά και νομικό τεχνικό επίπεδο, ε, να βοηθήσουν δηλαδή το Γενικό Εισαγγελέα και έχουμε αρχίσει ε, την πρώτη φάση ε, προσλήψεων για τους πραγματικούς υπαλλήλους, υπαλλήλου υπαλλήλους που θα στελεχώσουν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ελπίζουμε αυτή να είναι πλέον στη διάθεση του Εισαγγελέα το καλοκαίρι. μια άλλη διευκρινήση τώρα προ την κυρία Ζολή για το ρόλο του πάνελ επιλογής κατά την ανάλυση και την επιλογή των Ευρωπαίων εισαγγελέων. Έχω τους κανόνες εδώ μπροστά μου. Όντως το πάνελ έχει τη δυνατότητα, έχει λάβει την εντολή αν θέλετε, να απορρίψει μια υποψηφιότητα αφού θεωρεί ότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις προβλέπονται το άρθρο 16 του ε, ιδρυτικού κανονισμού. Υπάρχουν μια σειρά από απαιτήσει, θα θυμάστε, σχετικά με τις, τις, ε, τα προσόντα, την εμπειρία. Εάν το πάνελ κρίνει ότι δεν πληρώνται αυτέ οι προποθέσει, θα το διαβάσω στα αγγλικά τώρα μάλιστα, εφόσον λοιπόν οι υποψήφοι δεν πληρώνουν τι προποθέσει που αναφέρονται στο άρθρο 16, το πάνελ επιλογής μέσω τη, γραμματείας της, εγώ είμαι γραμ, γραμματεία αυτή τη στιγμή, θα στήσει από τα λόγο κράτη-μέλη να ορίσουν νέου υποψηφίου ίδιο αριθμό νέων υποψηφίων. Δηλαδή μπορεί να ζητήσει το πάνελ ε, από μια κρατημέλη να παρουσιάσει, από ένα να παρουσιάσει κάποιο νέο υποψήφιο. Τώρα για το δημοσιονομικό ζήτημα, όπω είπα, η εντύπωσή μα είναι ότι ο προπολογισμό που ψηφίστηκε για το 2019 αρκεί για την πρώτη φάση τη αρχική ε, λειτουργία. Θα δούμε από εκεί πέρα εάν θα χρειαστεί να επανέλθουμε στη συζήτηση ε, για τον προπολογισμό του 2020. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την προσοχή σας και την υποστήριξή σας και είμαστε στη διάθεσή σας να έρθουμε να σας ενημερώσουμε όσο χρειαστεί στο μέλλον. Ευχαριστώ. Okay, thank you. Ευχαριστώ. Να επαναλάβω για τους συναδέλφους ε, η ακρόαση θα γίνει στο δεύτερο μεσό του Φεβρουαρίου για το shortlist. μα είπε εδώ ο κύριος Σάλ, συζητήσαμε ήδη τη διαδικασία στην τελευταία συνεδρία συντονιστών. Ε, θα υπάρξει μια επικαιροποίηση όμως, θα μοιράσουμε στους συντονιστέ πριν από τη συνάντηση των συντονιστών ε, το σχετικό κείμενο και θα κάνουμε μια συζήτηση με βάση τα που ελέγχθησαν και σήμερα και αυτά που είπαν και οι συνάδελφοι, την ποιότητα δηλαδή των υποψηφίων και άλλα ζητήματα. Και βεβαίως στη συνέχεια θα αναφερθούμε, θα δώσουμε μια αναφορά εδώ στα μέλη. Ε, η συνείδηση των ζωνιστών θα λάβει χώρα μετά την συνεδρίαση τη σημερινή μας. Ευχαριστώ πολύ.